τις επεξηγήσεις ψήφου. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ για την έκθεση της κυρίας Άννας Γκόμες. Øh, Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Παρακαλώ λίγη ησυχία, αν μπορείτε. Παρακαλώ, όταν μιλάτε μεταξύ σας, ενοχλείτε αυτούς που κάνουν επεξηγήσεις ψήφου. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντική η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης. Θα πρέπει η Λιβύη να μην λειτουργεί ως χώρα ενδιάμεση για τους ε, λαθρομετανάστες από διάφορα σημεία του πλανήτη. Η Ευρώπη είναι ένας θαυμάσιος χώρος όπου καταφθάνουν οι πάντες. Και είναι όμως μια καταστροφή για όσους φτάνουν από χώρες φτωχές. Φτάνουν αυτά τα άτομα πάνφτωχα. Μιλάμε για άτομα που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Περνάνε λοιπόν μέσα από τη Λιβύη που γίνεται μια ενδιάμεση χώρα. Θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο λοιπόν στη σημερινή κατάσταση. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το συνεχές πέρασμα και η άφηξη των λαθρομεταναστών στα σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μουσκαρντίνη, θέλετε επεξήγηση ψήφου. Θα την κάνω γραπτός. Α, ευχαριστώ. μιλάμε για την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ε, θρησκευτικής ελευθερίας. Για κολλήνω Σαλβατόρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο αντισημιτισμός, ο αντισλαμισμός, αλλά και η εχθρότητα και η απέχθεια απέναντι στους χριστιανούς υπάρχουν σε, σε διαφορετικό βαθμό σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Ε, τα πρόσφατα γεγονότα που ορισμένα από αυτά ήταν αιματηρά με προβλήματα και επιθέσεις ε, σε χριστιανούς ε, στο, στην Ιγυρία, στο Πακιστάν και αλλού θα πρέπει να καταδικαστούν. Μιλάμε για παραγνώριση της θρησκευτική ελευθερίας. Ε, οι θρησκευτικές ελευθερίες θα πρέπει να εξασφαλιστούν και για τους χριστιανούς και για τους υπόλοιπους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε καν στη, στιγμή, στη σημερινή στιγμή οικονομικής κρίσης τη σημασία που έχουν αυτά τα γεγονότα. Μην ξεχνάμε ότι η Κομισιόν με 4 εκατομμύρια ευρώ υπερασπίστηκε την Ισλαμική, τη μουσουλμανική θρησκεία. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε χρησιμοποιήσει κάπου αλλού αυτά τα λεφτά. Είναι απίθανη αυτή η παρέμβαση Κομισιόν. Ευχαριστώ. Βεντινόρο αυτό που εγκρίναμε σήμερα είναι σημαντικό. Η θρησκευτική ελευθερία είναι η μητέρα όλων των ελευθεριών, αποτελεί τμήμα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που εκφράζονται και στην παγκόσμια διακήρυξη για τον άνθρωπο. Ε, υπάρχει το δικαίωμα ακόμα και να αλλάξει κανείς ελευθερία ή το δικαίωμα να εκφραστεί κανείς δημόσια και ιδιωτικά ε, για, την για την θρησκεία του και να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα όπως θέλει. Τα τελευταία, τις τελευταίες μέρες ε, είδαμε γεγονότα εναντίον θρησκευτικών μειονοτήτων, κυρίως χριστιανικών μειονοτήτων, σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Ε, έτσι αμφισβητείται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας σήμερα. Υπάρχει ε, μυσαλλοδοξία, ε, η οποία χρησιμοποιείται για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Σε αυτό το κλίμα αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν στην πραγματικότητα σοπαίνουν σήμερα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα τμήμα των ανησυχιών που εκφράστηκαν μπορώ και εγώ να το συμμεριστώ. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει εδώ πέρα στην έκθεση δηλαδή το εκτιμώντας 7 για τις τουρκικές αρχές και το τι κάνουν στη Βόρεια Κύπρο. Μιλάμε για παράνομα κατεχόμενη χ υπό τουρκική κατοχή, οι οποίοι οι Τούρκοι ταυτόχρονα διαπραγματεύονται μαζί μας για έντοξη. Οι δε Ελληνοκύπροι που θέλουν να επιστρέψουν ε, στο σπίτι τους και να λειτουργήσουν τις ε, εκκλησίες, τα μοναστήρια κτλ. δεν μπορούν να το κάνουν, δεν μπορούν καν να τις αναστηλώσουν. Δεν μιλάμε βεβαίως για τις ιδιοκτησίες τους και τα Αυτά ζούμε στη Βόρεια Κύπρο. Είναι μια διάκριση και καταπίεση των χριστιανών που γίνεται από μια χώρα που θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να συστήσουμε να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μέχρι να λυθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη από τις ρίζες της έχει μια συγκεκριμένη υποχρέωση να προστατεύσει όλους τους χριστιανούς ανά τον κόσμο. Το ψήφισμα αυτό αποτελεί φυσικά έκφραση ακριβώς του γεγονότος αυτού και πρέπει να το στηρίξουμε. Από την άλλη πλευρά όμως η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε ενέργειες που και στο μέλλον θα προστατεύουν όλους τους χριστιανούς ανά τον κόσμο και δεν θα οδηγούν σε παρόμοιες τραγωδίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσφατα, σε διάφορες χώρες όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, υπήρξαν ε, διώξεις ε, καθολικών. Δεν μπορούμε να σταθούμε διάφοροι. Το πρόβλημα της ε, αναγνώρισης της θρησκευτική ελευθερίας είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό υποστηρίζω τη δήλωση του Προέδρου Μπούζεκ που μίλησε εναντίον αυτών των δράσεων και θα ήθελα να υποστηρίξω και όλες τις δράσεις για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των θρησκευτικών μειονοτήτων εκεί όπου παραβιάζονται τα δικαιώματά τους στην έκθεση του 2009 για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτή την προστασία ανά τον κόσμο και ζητήσαμε να υπάρξει ένας ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το σημερινό ψήφισμα είναι ένα θαυμάσιο βήμα, πρώτο βήμα για την μάχη αυτή. Ο κύριος Αντρέι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος. Ήμουν συνεισηγητής και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άστον για την αντίδρασή της στη δίωξη χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Θυμόμαστε και τους Ιρακινούς επισκόπους και την αντίδρασή τους στη δίωξη των χριστιανών του Ιράκ. Θα ήθελα να πω πως σε λίγους μήνες θα έχουμε την αγιοποίηση του Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου, του Πάπα. Και μακαριοποίηση. Και μπορούμε βεβαίω να λύσουμε από τα διδάγματά του, καθώς πάντα πέρα από τις εκκλησίες ανέφερε και τα τζαμιά και τις συναγωγές. Αυτό είναι το καθήκον μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και βεβαίως να υποστηρίξουμε αυτούς που έξαν πολλά λόγω Κέλαμ. Κέλαμ. Έχει το λόγο. Ε, Πρόεδρο, πρόεδρε, υπερψήφισα το ιστορικό αυτό ψήφισμα και ήμουν και εγώ συντάκτης του. Υπάρχουν δύο σημαντικά μηνύματα λοιπόν εδώ πέρα προς την ύπατη εκπρόσωπο και προς την Κομισιόν που θα πρέπει να εκτελεστούν το συντομότερο δυνατόν. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν πρέπει να αναπτύξει επιγόντως μια στρατηγική της Ένωσης για την επιβολή του δικαιώματος της θρησκευτική ελευθερίας συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά κρατών που δεν προστατεύουν θρησκευτικές μειονότητες. Και δεύτερον, η Κομισιόν πρέπει να αναπτύξει ένα μόνιμο σύστημα εντός της Διευθύνσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να παρακολουθεί κυβερνητικούς περιορισμούς στη θρησκευτική ελευθερία και να δίνει λόγο κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μουσκαρδίνη. Πρόεδρε, η θρησκευτική ελευθερία είναι βασική αξία του πολιτισμού μας. Χωρίς ε, την, αυτή η δημοκρατία είναι ακροτηριασμένη και νομίζω ότι αρνείται στον άνθρωπο την, την αξιοπρέπειά του. Αυτό συμβαίνει ε, σε διάφορα τμήματα του κόσμου όπου ρηξικέλευθες και ε, εξτρεμιστικές τάσεις ε, σκοτώνουν χριστιανούς. Αυτοί είναι μάρτυρες. Η έλλειψη ανεκτικότητας υπάρχει μέσα σε αυτή την κουλτούρα την φονταμενταλιστική και οποιαδήποτε έκφανση άρνησης της θρησκευτική ελευθερίας ε, νομίζω ότι πληγώνει την αξιοπρέπεια παντού και νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις ε, σφαγές των χριστιανών. Ε, οι κόπτες ας πούμε της Αιγύπτου αλλά και οι χριστιανοί του Ιράκ κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Είναι παρόντες σε αυτές τις περιοχές για αιώνες. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούζεκ που αποτελεί φως με τις δηλώσεις του για όλους τους χριστιανούς που είναι θύματα του Ισλαμικού ε, φονταμενταλισμού. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε ε, νομίζω το λίκνο της ελευθερίας για την ανθρωπότητα. Χωρίς αυτή την ελευθερία δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν μια σειρά από αξίες. Μια σειρά από αξίες καταπατώνται. Και εγώ ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, ε, γιατί το θέμα της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών ανά τον κόσμο είναι σήμερα πολύ επίκαιρο. Είναι πολύ ανησυχητικό το 2011 ότι κάποιος ε, διώκεται μόνο και μόνο λόγω της πίσης του. Το άρθρο 10 της ε, Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει τέτοιες ερμηνείες. Λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκευτικής συνείδησης. Ε, τις τελευταίες οι θρησκευτικέ επιθέσεις είναι σημάδι ότι είναι και η ώρα όλες οι κυβερνήσει, παρά τις δυσκολίε και τις απειλές να υιοθετήσουν μέτρα για την προστασία όλων των θρησκευτικών ελευθεριών. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να υπάρξει ένας ε, διάλογος μεταξύ των θρησκειών, μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά κυρίω. Ε, μεταξύ αυτών ε, όπου δεν εξασφαλίζουν την ε, θρησκευτική ελευθερία κυρίως. Θα πρέπει αυτή η θρησκευτική ελευθερία να εξασφαλιστεί παντού χωρίς εξαιρέσεις. Ευχαριστώ την κύριο Τσούλη. ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καλό ψήφισμα. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ανεξιθρησκεία στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τις ρίζες μας. Τις ισχυανικέ παραδόσεις αλλά και τις ευρωπαϊκές αξίες οι οποίες είναι βασισμένες στις ρίζες αυτές που ανέφερα. Τα γεγονότα που συνέβησαν με τους κόπτες στην Αίγυπτο μας κάνουν να δούμε ότι και οι χριστιανοί χρειάζονται ειδική προστασία σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αίγυπτο. Παρόμοια περιστατικά έχουμε στην Τουρκία, στη Συρία, αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τέτοια κρούσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκονται. και νομίζω ότι φοβούμαστε τον Ισλαμισμό, αλλά έχουμε απεμπολίσει τι δικέ μα αξίε. Δεν είναι σωστό ο τρόπο αυτό. Χρειαζόμαστε διάλογο, χρειαζόμαστε θρησκευτική ελευθερία και πρέπει όμω να εμείνουμε και στι βασικέ μα αξίε, που είναι τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χριστιανικές αξίες και πρέπει να παραμείνουμε, να εμείνουμε σε αυτά γιατί είναι και το τμήμα της ταυτότητάς μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλέης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα το ψήφισμα αυτό και χαίρομαι που εγκρίθηκε. Αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες για την διατύπωση που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα δίνει την εντύπωση πως τα μεγαλύτερα προβλήματα των χριστιανών είναι στις μουσουλμανικές χώρες. Αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα με τη θρησκευτική ελευθερία. Αλλά τι κάνουμε εδώ πέρα. Φέρνουμε τα μεμονωμένα προβλήματα και περιστατικά στην Ευρώπη σε ίδια μοίρα με τα διαρθρωτικά και θεσμικά προβλήματα διάκρισης των ε, χριστιανών στις μουσουλμανικές χώρες. Δηλαδή εκεί πέρα είναι επίσημη πολιτική του κράτους. Σκεφτείτε το πως είναι αδύνατο να ανακαινιστούν εκκλησίες στην Τουρκία παραδείγματος χάρη, δίωξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου της ε, Κωνσταντινούπολης, να μην μιλήσουμε για το τι γίνεται από τις δυνάμεις κατοχής στην Κύπρο. Αυτά είναι σκάνδαλα. Ευχαριστώ. Uh, Κέλλη. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούζεκ για την, τον ηγετικό ρόλο που παίζει. Ε, σήμερα θυμόμαστε, ξανθυμόμαστε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου οι, διώκονται πάλι οι χριστιανοί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να κάνει και αυτή ό,τι μπορεί, να παίξει το ρόλο της. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη θρησκευτική ελευθερία για τις διάφορες θρησκευτικέ ομάδες, ε, αλλά και στις χώρες που κάνουν αίτηση ένταξης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ίδιο. Αυτά τα ψηφίσματα πέρασαν και πέρασαν ομόφωνα. Χαίρομαι γι' αυτό. Ο κύριος, ευχαριστώ τον κύριο Κέλλη. Uh, Θα σας ε, μιλήσω. Εγώ ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση στη Λευκορωσία ή ε, δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Μετά, ο κύριος Τσαρνέσκι. Πρέγω. The same. On... Δεν είσαστε εδώ, κύριε Τσαρνέσκι. Θα μιλήσετε ή όχι. Grazie, Presidente. Uh, proszę Państwa, Ευχαριστώ. Αυτό το ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι το πρώτο και ψηφίζεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Ξέρουμε τα προβλήματα των χριστιανών στο Ιράκ, ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αίγυπτο. Τα τελευταία χρόνια δεν συνέβαιναν αυτά που συνέβησαν τώρα. Ξέραμε για μεμονωμένες περιπτώσεις ε, Ξέρουμε για δολοφονίες χριστιανών, ξέρουμε ότι στη Συρία, Τουρκία και στο Πακιστάν δολοφονούνταν και χριστιανοί ιερείς. Ξέρουμε τι συμβαίνουν σε κάποιες αφρικανικές χώρες, ε, όπου ζουν κυρίως μουσουλμανικές ε, πλειοψηφίες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμω είναι η σιωπή του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του κ. Μπαρόζου. Ε, επί μία εβδομάδα δεν είπε τίποτα, ενώ πολλοί α, πρωθυπουργοί και κράτη-μέλη ε, άσκησαν πίεση, εν πάση περιπτώσει κάναν κάποιε δηλώσει. Εκείνο όμω δεν είπε τίποτα. Τήρησε σιγή χθείο. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στι δηλώσει για την έκθεση για την κατάσταση στην Λευκορωσία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που γνωρίζουμε εδώ μέσα το ότι διολυσθένει προς τον αυταρχισμό η Λευκορωσία σε ένα σύστημα που το είχαμε ξεπεράσει πριν από 20 χρόνια. Όμως το ψήφισμα αυτό μπορεί να προκαλέσει ίσως κάποια αυτοκριτική σε κάποιους συναδέλφους. Δηλαδή ας αναλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας απαράτσικ της Ένωσης θα δει πολλές ομοιότητες. Βλέπω ε, δεν μας κυβερνά ερετός πρόεδρος, αλλά ένα πολίτμηρο 27 μελών που λέγεται Κομισιόν. Βλέπετε ένα κοινοβούλιο που μόνο τυπικά εγκρίνει τα πράγματα. Θα νοσταλγούσε. Θα νοσταλγούσε επίσης και τα πενταετή προγράμματα. Θα τα βλέπε εδώ πέρα. Θα βλέπε επίσης τον στόλο των ε, λιμουζινών ε, και ειδικών μαγαζιών για την νομεκλατούρα. Επίσης θα έβλεπε αυτό το οποίο ο είπε το σύστημα τη λανθασμένη συνείδηση. Ο κόσμο ψηφίζει και δεν καταλαβαίνει τα συμφέροντά του. Είναι τρομακτικό αυτό και θυμίζει την φάρμα των ζώων που στο τέλος κοιτάμε ανθρώπου και γουρούνια και δεν μπορούμε να πούμε τον ένα από τον άλλον. Ευχαριστώ. υπό. Ευχαριστώ πολύ. Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό Νομίζω ότι θα πρέπει να υπαγρυπνά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανατολή. Επίσης πρέπει να δούμε συγκεκριμένα και τα προβλήματα της νεολαίας. Ε, οι νέοι στη Λευκορωσία και οι οργανώσεις της νεολαίας δεν έχουν ελευθερία κινήσεων. Στην Ευρώπη εδώ και χρόνια έχουμε την παράδοση να διοργανώνουμε κάποιες ε, εκδηλώσεις, κάποιες διαδηλώσεις κατά της παραβίασης των δικαιωμάτων. Ελπίζω η Λευκορώσοι να μην βλέπουν εμάς άφωνους, μουγκούς, αλλά να υποστηρίξουμε και εμείς τις αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίσενιν από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, θα μιλήσει για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών υποστήριξε το ψήφισμα. Πιστεύουμε ότι θα στείλει ένα έντονο μήνυμα και στις ε, λευκορωσικές αρχές και στην κοινωνία των πολιτών και στα ΜΜΕ που όλοι μάχονται για την δημοκρατική ανάπτυξη της ε, χώρας. Τα μέτρα που περιλαμβάνει το ψήφισμα θα αναλυθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και ταχεία δράση θα αναλυθεί για να υπάρξουν και αποτελέσματα. Υπάρχει αυτή η τελετή ε, που έχει προγραμματιστεί για αύριο που όμως δεν θα αφημώσει τις ανησυχίες για τον τρόπο που εξελέγει ε, ο του Κασέγκο. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί και πολιτικές για να επηρεάσουμε την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ε, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής όμως είχε μέτρια αποτελέσματα. Ίσως θα πρέπει να δούμε νέους τρόπους, να βρούμε και νέες μεθόδους. Ε, ίσως χρειάζονται νέοι μηχανισμοί. Το ψήφισμα υπονοεί ότι υπάρχει κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί. Συντονισμός των μέτρων και της τάσης μας προς την ε, Λευκορωσία με αυτή των γειτόνων που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας που είναι στρατηγικός εταίρος και της Ουκρανίας που είναι τμήμα της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Μια κοινή συντονισμένη δράση μπορεί να πετύχει τουλάχιστον τη δημιουργία ενός καταλληλότερου πολιτικά περιβάλλοντος ε, που θα καταστήσει δυνατόν την διενέργεια ε, πραγματικών και ανώθευτων εκλογών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ε, τις δυνατότητες που έχει. Σήμερα αποφασίσαμε να στείλουμε μια αντιπροσωπεία στη Λευκορωσία. Νομίζω ότι θα είναι μια δοκιμασία για την ηγεσία της Λευκορωσίας αν δώσει πρόσβαση σε αυτή την αντιπροσωπεία και αν της επιτρέψει να δει ε, εκ του την κατάσταση. Ο κύριος Σόνικ Μπόγκοσλαβ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω πόσο με εξοργίζει αυτή η σύγκρουση η σύγκριση με τη Λευκορωσία έχουν ακουστεί ανοησίες πάρα πολύ δυσάρεστες και μάλιστα χειροκρότησαν και οι συναδελφοί μου από την ομάδα των συντηρητικών κάποιες από αυτές τις ανοησίες. Το καθεστώς του Λουκασέκο πρέπει να απομονωθεί. Αυτό που νομίζαμε ότι θα γίνει, δηλαδή ότι η πολιτική του θα γίνει σιγά σιγά δημοκρατική, έδειξε ότι αυταπατηθήκαμε. Θα πρέπει να του επιβληθούν βαθιές κυρώσεις, γιατί είναι ε, μια χώρα πολύ κοντά στην Ευρώπη και σε σχέση με τη χώρα αυτή θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει και προσδοκίες. Θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την ελευθεροτυπία και την ελευθερία των τηλεοπτικών σταθμών που ενημερώνουν τον λαό της χώρας. Πιέλανα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα γεγονότα στη Λευκορωσία σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές έχουν να ακόμα μια φορά την κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Για μια ακόμα φορά ο πρόεδρος Λουκασένκο χρησιμοποίησε βία εναντίον των αντιφρονούντων. Ε, είναι στη χειρότερη φάση της δικτατορίας, τους, ε, δικτατορίας του. Έχει ε, συλλάβει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και παραβιάζει σαφώς τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τάσεις του. θα Γι' αυτό ακριβώς είμαι υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάει άμεση απελευθέρωση των ε, κρατουμένων. Καταδικάζω τις ε, ε, δικτατορικές πρακτικές του καθεστώτος Λουκασέγκου και πιστεύω ότι η πίεση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μειώσει την καταστολή εναντίον των λευκορώσων πολιτών. Παράλληλα, Είμαι υπέρ όλων των δράσεων, υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών. Ε, υποτροφίες για ερευνητές και συγχρηματοδότηση των ανεξάρτητων ΜΜΕ. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η Λευκορωσία είναι πραγματικά ντροπή για εμάς ε, στην Ευρώπη. Είναι η τελευταία κομμουνιστική δικτατορία και πρέπει βεβαίως να ασκήσουμε κριτική. Αλλά ε, ξέρετε, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Γι' αυτό πρέπει να δούμε λίγο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σκοπιά της Λευκορωσίας. Υπάρχει μια κομισιόν άνθρωποι που δεν έχουν καμία εντολή από τον ε, λαό. Δεν έχουν ε, εκλεγεί αλλά κάνουν προτάσεις οι οποίες γίνονται νόμοι και βεβαίως ε, έχουν πολύ σημαντικές ε, συνέπειες στα κράτη-μέλη. Μετά οι δικαστές είναι απομακρυσμένοι από όλους τους υπόλοιπους, το ίδιο και εδώ μέσα στο κοινοβούλιο οι περισσότεροι αισθάνονται μια χαρούλα εδώ μέσα στο γυάλινο αυτό παλάτι που καθόμαστε. Δεν έχουν πλέον επαφή με την ε, πραγματικότητα και τις ανησυχίες ε, των ε, λαών της Ευρώπης. Αν τα δει κανείς λοιπόν αυτά από τη σκοπιά της Λευκορωσίας μπορεί να πει πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δικτατορία που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Κύριος Τσαρνέσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε υποστήριξα αυτό το ψήφισμα, γνωρίζοντας ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι πολύ ιδιαίτερη. Εδώ ασχολούμαστε με μια ανεξέλεγκτη βία εναντίον ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό προκαλείται από μια απαράδεκτη πολιτική κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικές που δεν τις έχουν σκεφτεί και χωνέψει καλά, οι οποίες νομιμοποιούν τον κύριο Λουκασέγκο. Ε, με τις επισκέψεις στη Λιθουανία και στην Ιταλία πραγματικά νομιμοποιείται το, καθεστώ του, το καθεστώς του. Ε, και με επισκέψεις στην Γερμανία και στην Πολωνία. Ήταν περιττές αυτές οι επισκέψεις. Θα πρέπει να Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στην Λευκορωσία. Μάλιστα, πάμε τώρα στην έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Κόσλικ. Ο κύριος Κόσλικ έχει το λόγο. Vážený pán prezident, kolegovia, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η εμπειρία από τα κράτη-μέλη δείχνει πως ε, έξι χρόνια μετά τον κανονισμό 1-2003 του Συμβουλίου δεν υπάρχει αλλαγή όσον αφορά τους κανόνες του ανταγωνισμού. Τα εθνικά δικαστήρια απευθύνονται στο ΔΕΚ με ε, ερωτήματα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις του ανταγωνισμού, ούτε καν με προδικαστικά ερωτήματα. Και εκεί πέρα σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν έχει χρησιμοποιήσει και η Κομισιόν το δικαίωμα να παρέμβει ως αμήκους κούριε. Το πρόβλημα λοιπόν ε, εδώ πέρα είναι η εφαρμογή στην πράξη. Γι' αυτό απευθύνομαι προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει μέτρα για να επιτευχθούν αυτοί οι ε, στόχοι, για να υπάρχει ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσσερμιτ ξανά. Er Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, υπάρχει αμφιβολία. Η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη είναι υποπίεση. Υπάρχει θέληση να αλλάξουμε κάτι στα κράτη-μέλη. Ναι, εντάξει, δημιουργήσαμε το κοινό νόμισμα που καταστρέφει αυτή τη στιγμή ολόκληρη την Νότια Ευρώπη βεβαίως. Και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν ε, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε την Ινδία, την Κίνα, τη Λατινική Αμερική. Ε, είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε. Υπάρχει μια πρωτοβουλία, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Άλλη καταστροφή εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και αυτό δείχνει πόσο αναποτελεσματική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χανόμαστε στα τεχνικά. Ε, απλά είναι τα πράγματα. Πράγματα που χρειαζόμαστε δηλαδή και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά. Οπότε ποια είναι αυτή η συνεργασία τελικά. Πρέπει να δούμε ποια είναι η βάση. Πρέντα. Παρέμβω για το θέμα της Λευκορωσίας, κύριε Πρόεδρε. Για τη Λευκορωσία τελειώσαν οι επεξηγήσεις ψήφου. Έπρεπε να είχατε γραφτεί πριν. Μπορείτε όμως να μας δώσετε την επεξηγήσή σας γραπτός όμως. Επαναλαμβάνω, για τη Λευκορωσία τις έχουμε τελειώσει τις επεξηγήσεις ψήφου. Αν θέλετε μπορείτε να μας κάνετε την επεξήγησή σας γραπτός. Αλλιώς έπρεπε να είχατε γραφτεί πριν. Ακαπίτο. Με καταλάβατε. Με καταλάβατε. Ε, μπορώ να το πω τώρα. Δεν μπορείτε τώρα να κάνετε την επεξήγησή σας πριν έπρεπε να την είχατε κάνει, όταν γινόταν οι άλλε επεξηγήσει για τη Λευκορωσία. Εσεί όμω δεν μα ζητήσατε το λόγο, άρα δεν σα έδωσα το λόγο. Μπορείτε όμω τώρα να μα στείλετε το κείμενό σα γραπτό. Καταλάβατε τώρα. Μπράβο. Στείλτε μα το κείμενό σα γραπτό. Κυρία Μουσκαρντίνη. Πρόεδρε, ε, εκτιμώ την ευελιξία της ε, Κομισιόν για την, ε, τους, του ορισμού για τι κρατικέ ενισχύσει. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση λεπτομερής για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, ούτω ώστε να υπάρχουν οι ίδιε συνθήκε ανταγωνισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την πρόσκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζε επιστρέφουν τι κρατικέ ενισχύσει που λάβανε, οι οποίε ήταν τεράστιε, για να υπάρξει ίση ίσως ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Ε, θεωρούν ορισμένοι ότι αυτές οι ενισχύσεις, οι τεράστιες με τα λεφτά των φορολογουμένων, ε, ήταν εξωφρενικές, αλλά χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δημόσιο χρήμα για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη. Ε, η αποταμίευση όμως των μικρομεσαίων δεν θα πρέπει στην πραγματικότητα να είναι ε, τροφή για τους τραπεζίτες. Ε, χαίρομαι για την, το άνοιγμα που υπάρχει ε, υπέρ κοινών ε, με σκοπό να αναπτυχθεί η ανανεώσιμη ενέργεια. Ευχαριστώ κυρία Μουσκαρδίνη. Ο κύριος Κέλλη. Ε, Κύριε Πρόεδρε, με χαρά υποστήριξα αυτή την, αυτό το ψήφισμα γιατί πρωταρχικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχει ε, να διασφαλίσει τον θεμητό ανταγωνισμό κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Υπάρχει υπόψη ότι υπάρχει εκμετάλλευση των αγορών και στη χώρα μου υπάρχει ανησυχία γιατί έχουμε ε, αύξηση των τιμών ε, του πετρελαίου και άλλων που θα επηρεάσουν και τις γεωργικές τιμές. Υπάρχει η υποψία ότι υπάρχει ένα καρτέλ ιδίω σε ό,τι αφορά τη μείωση των ε, τιμών των ε, βοηδών. Και πάρα πολύ πρόσφατα είδαμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά εταιριών τηλεπικοινωνιών για τις κλήσεις περιαγωγής και τις χρεώσεις τους. Πρέπει να είμαστε συνεχώς λοιπόν σε παγρύπνηση και να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε άμεση δράση σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένα κρούσμα θέμη του ανταγωνισμού. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση που έχει συνταχθεί από έναν έμπειρο συνάδελφο. Και πρέπει να πούμε ανοιχτά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει περισσότερη διαφάνεια και ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε αυτά. Αυτό, αυτά μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Ευρώπης σε, μια, σε ένα τομέα που είμαστε πίσω. Πρέπει να πούμε την αλήθεια όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία. Τα ψηφίσματα μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό χρειάζονται. Πάμε τώρα στο ψήφισμα για τη βιώσιμη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον απότατο βορρά. Ο κ. Τάκουλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μίκαελ Γκάλερ γιατί είναι θαυμάσια αυτή η έκθεση. Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των υπερβόρειων περιοχών της Υπήρου μας. Εγώ παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία και τα ιδιαίτερα ζητήματα του κλίματος, τα οικονομικά ζητήματα, ε, η ζωή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί, η γεωργία, η εκτροφή των ταράνδων, όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Επίσης έχουμε το θέμα των Σάμι, των γηγενών πληθυσμών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάλερ, ο οποίος ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας ε, γίνεται κέντρο ε, πληροφοριών για τον αρκτικό κύκλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που οι Φιλανδοί ξεπέρασαν τις αγκυλώσεις τους ε, και αγκαλιάζουν τώρα τον Βορρά. Η έκθεση Γκάλερ ήταν θαυμάσια και τον ευχαριστώ τον κύριο Γκάλερ. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εύξηνο πόντο. Ο κύριος Βίσενιν από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για δύο λεπτά. Κύριε Βίσενιν. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου πιστεύει ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εύξηνο πόντο είναι πολύ σημαντική και έρχεται και στην κατάλληλη χρονική στιγμή διότι ουσιαστικά ε, εξισορροπεί τα όσα έχουν ε, επιτευχθεί μέχρι τώρα και κάνει κάποιε προτάσεις για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη στο μέλλον. Νομίζουμε ότι η πολιτική συνεργασία με εταίρους ε, που έχουν διαφορετικά επίπεδα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεν δύσκολο εγχείρημα, αλλά όχι ακατόρθωτο. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τι προσπάθειέ μα σε πολιτικό επίπεδο. Τρει χώρε είναι μέλη τη Ένωση. Ένα είναι στρατηγικό εταίρο, άλλε χώρε είναι μέλη στρατική σύνθεση και η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα. Μιλάω για τι παρεξήνιε χώρε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη βούληση. Γιατί στερούμαστε ένα σημαντικό δυναμικό μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή δηλαδή η συνέργεια των εύξενο πόντο που από την αρχή θεωρήθηκε ως μια φιλόδοξη πρωτοβουλία θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε μια πραγματική στρατηγική. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συνεργασίας που μπορούν με κάποιες προσαρμογές να αξιοποιηθούν όπως είναι η στρατηγική για τη Βαλτική, ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασία συγκεκριμένα. Νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν διάφορα βήματα και να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Δεν έλειψαν υπόψη όλε μα οι προτάσει. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο τη στρατηγική στρατηγικής τη πολιτική γειτονία, Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο του πώ μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ στρατηγική για τον ξενοπόντο και ανατολική εταιρική σχέση εφόσον οι περισσότερες χώρες ε, ε, έχουν ε, προσχωρήσει στην Ανατολική Εταιρική Σχέση πλην Λευκορωσίας. Και σε υπουργικό και σε βουλευτικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε περισσότερο τη στρατηγική για τον Εύξηνο Πότο με τη στρατηγική για το Δούναβι με αποτέλεσμα μια στρατηγική η οποία θα έχει και ξεχωριστό κονδύλιο του προπολογισμού στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ, Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία για στρατηγική που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα Αγκουρεάνου πρέπει να υποστηριχθεί και η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η ανατολική εταιρική σχέση με τη Ρωσία και η διαπραγματεύσεις για ένταξη δικαιολογούν την πολιτική σημασία αυτής της περιοχής για την Ένωση. Είναι μια σημαντική περιοχή για τη διέλευση ενεργειακών πόρων και από μελλοντικών έργων όπως ο Ναμπούκο που είναι πάρα πολύ σημαντικός για να αλλάξουμε προμηθευτές φυσικού αερίου. Επίσης, συμφωνώ με τον εισηγητή, τον οποίο θέλω να συγχαρώ, ε, στο ότι πρέπει να λάβουν υπόψη όλε οι χώρε, όχι μόνο τι μεγάλε χώρε περιοχή και βέβαια η στρατηγική αυτή να είναι συμβατή με άλλε όπω π.χ. η στρατηγική τη Μεσογείου. Ευχαριστώ, Σάρους. 2007-ben, mikor Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz, a Fekete-tenger részben az Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε πως όταν μπήκαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον άρχισε να βρέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Μαύρη Θάλασσα και είναι πολύ στρατηγικής σημασίας ο χώρος αυτός για την Ένωση. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια οικονομική στρατηγική και να αποκτήσει και μια γραμμή στον προϋπολογισμό. Η στρατηγική της Ένωσης ε, πρέπει να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε διάφορες πηγές και δρόμους και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέρμιναλ υγρών ε, καυσίμων. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ασφαλή ενεργειακή παροχή στην Ένωση Νομπούκο και ο διευρωπαϊκός αγωγός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το και το υποστήριξα. Τελειώσαμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και για τη Λευκορωσία, ήθελα να κάνω μια επεξήγηση ψήφου για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εύξηνο πόντο. Καταρχάς, η ιδέα του κύριου Ουγγουρεάνου να ετοιμάσει έκθεση για αυτό το θέμα ήταν πολύ καλή. Επαναλαμβάνω ότι η ιδέα του κύριου Ουγγουρεάνου να συντάξει αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας ε, έρχεται την κατάλληλη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενδυναμώσει την πολιτική της με στρατηγικές για, για τον εύξηνο πόντο όπως αντίστοιχες με αυτές της Βαλτικής και του Δούναβη. Ε, χαίρομαι που οι τροπολογίες μου υπάρχουν στο κείμενο της τροπολογίας. Ε, μιλάω για ένα δίκτυο που θα πρέπει να δημιουργήσει στην περιοχή. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, προγράμματα ε, μεταξύ για το διάλογο μεταξύ των θρησκειών και τον πολιτισμό αλλά να δημιουργήσουμε και ένα πανεπιστήμιο ε, στον εύξηνο πόντο. Νομίζω ότι η ανάπτυξη επίσης της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να ε, επηρεάσει θετικά και τις πολιτικές εξελίξεις. Ε, επίσης, προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμογή της σύμβασης της Μαύρης Θάλασσας κατά της ρήπανσης, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και ελπίζω το Συμβούλιο να δώσει σημασία σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Την επόμενη φορά κύριε Πρέντα σας παρακαλώ να καταγράψετε, να σημειώσετε και να ζητήσετε ε, να μιλήσετε. Ε, όχι, ζήτησα να μιλήσω. Όχι, δεν ζητήσατε να μιλήσετε. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτή τη φορά, αλλά την επόμενη φορά σα παρακαλώ να ζητήσετε εκ των προτέρων να μιλήσετε. Εντάξει, καλή όρεξη. Σταματάμε τώρα τη συνεδρίαση μέχρι τι 3 η ώρα.